Ευχαριστώ συνάδελφοι για την κατανόησή σας. Ε, περιμέναμε να τελειώσει η διάσκεψη των Πρόεδρων, σχεδόν έχει τελειώσει. Πριν αρχίσουν οι ψηφοφορίες έχω δει διαδικαστικά από την κυρία